Dichiaro επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση τη Ολομέλεια που διακόπη στι 2 Μαρτίου του 2017. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου